αυτού Μακάλιστερ από το Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Η Ταλακριτική Ευρώπη επλήγει από πλημμύρες για τη Σερβία, την Βοσνία Ζεγοβίνη, την οποία επισκέφτηκα τη Σερβία πριν από λίγες εβδομάδες και πραγματικά οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελαφρύνουν τα πλήγματα από τις περσινές πλημμύρες επισκέφθηκα την πόλη της Σιγάινα που επλήγει πολύ σοβαρά πήγαμε σε ένα νηπιαγωγείο και σε κτίρια τα οποία χτίστηκαν και ανακαινίστηκαν με, τους, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είδαμε ότι οι προσπάθειές μας εκεί πραγματικά είμαστε ο κυριότερος ε, δωρητής στην περιοχή αυτή και χάρη σε αυτήν την βοήθεια μπόρεσαν κτίρια, σπίτια να χτιστούν, να ανακαινιστούν. Σήμερα όμως Σήμερα πρέπει να γίνουν έργα προληπτικά αυτών των καιρικών φαινομένων. 90 19 συγγνώμη, εκατομμύρια θα διατεθούν για αυτά τα έργα και θεωρώ πραγματικά ότι θα πρέπει όλοι μαζί να συνεισφέρουμε έτσι ώστε στο μέλλον να αποφευχθούν παρόμοιες πλημμύρες και καταστροφές. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Η, κυρία Αλέσια Μαρία Μόσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες εβδομάδες τα στατιστικά στοιχεία για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης ε, για τα ε, ε, φροντίδα για βρέφη. Μόνο σε επτά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει καλή ποιότητα. Οι υπηρεσίες ποιότητας ε, χαρακτηρίζονται από έλλειψη πόρων. Αυτό συνεπάγεται δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων και δημιουργεί χάσμα μεταξύ των φίλων, διότι οι γυναίκε είναι αυτέ που πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά λόγω απουσίας υπηρεσιών. Γι' αυτό ζητάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει, να εγγυηθεί σε όλους του τους πολίτες ε, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους μαζί με άλλα μέτρα που θα συμβάλλουν στη μείωση οποιασδήποτε μορφής διακριτική μεταχείρισης όπως ενημέρωση προς όλους ε, για τις γονικές άδειες και ε, πρόθεση του smart working που θα επιτρέψουν όχι μόνο στις γυναίκες αλλά σε όλους τους εργαζομένους να συμφιλώσουν καλύτερα την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φωνστόρκ. Ja, morgen wird in diesem Ευχαριστώ. Αύριο για άλλη μια φορά εδώ θα μιλήσουμε για την άμβλωση. Είναι ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται και κάθε φορά λέμε ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα σε καμία περίπτωση της Ευρώπης και δεν θέλω να δαπανώνται χρήματα για να συζητούνται εδώ θέματα που είναι προφανές ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρώπης. Και αναφέρομαι εδώ στην έκθεση Ταραμπέλα. Στην Γερμανία η άμβλωση τιμωρείται μέχρι και με τρία χρόνια φυλάκιση. Και εδώ βλέπουμε η έκθεση Ταραμπέλα να ζητάει την απελευθέρωση των αμβλώσεων. Αναφέρεται στην άμβλωση σαν ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Εμείς θέλουμε να επικαλεστούμε εδώ κάποια άλλα θεμελιδόλη δικαιώματα όπως το δικαίωμα της ζωής, την προστασία στην ζωή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Ιβάν Γιάκοψη από την Άλντε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μία από τις μεγάλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η περιβαλλοντική και η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτά ε, λοιπόν αφορούν ιδιαίτερα στην πολιτική που ακολουθούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Αφορούν το στόχο που έχουμε για λιγότερη εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τον άνθρακα. Ωστόσο και δυστυχώς πολύ γρήγορα θα καταλάβουμε, θα δούμε ε, κατασκευή στην Ίστρια ε, ρηπογόνου εργοστασίου. Αυτό δεν πρόκειται καθόλου να προστατεύσει το περιβάλλον. Είναι μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Και ξέρετε, κοντά σε αυτές τις εγκαταστάσεις υπάρχει ένα έργο που έχει συγχρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ΚΕΡΚ. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου για να λειτουργήσουν με φυσικό αέριο και όχι με ε, άνθρακα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροντρίγκεθ, παρακαλώ. Sí. Gracias, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, μία μέρα μετά τον εορτασμό της 8ης της ε, Μαρτίου, ε, διεθνούς ημέρας ε, των γυναικών, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τον τρόπο με τον οποίο διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικές λιτότητας πλήττουν πολύ περισσότερο τις γυναίκες. Οι περικοπές πλήττουν ιδιαίτερως γυναικείους τομείς όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η δημόσιο, ο δημόσιος τομέας. Η λιτότητα εξαφανίζει τα μέτρα στήριξης και συμφιλίωσης και έτσι η γυναίκα αναλαμβάνει ακόμα περισσότερο το άχθος των οικιακών εργασιών, της φροντίδας των ηλικιωμένων, τη φροντίδα των παιδιών μαζί με τη δουλειά της. Οι περικοπές ε, ε, πλήττουν τις πολιτικές μας για την καταπολέμηση της ανδρικής βίας. Η μισθή είναι πολύ χαμηλότερη στις γυναίκες, η μισθή των γυναικών. Στη Γαλλικία οι γυναίκες πληρώνονται 24% λιγότερο από ότι οι άνδρες και Συνεχίζουμε οι γυναίκες να μην αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά μας δικαιώματα εντός οικογένειας. Η φτώχεια έχει θηλυκό πρόσωπο. Το 70% όσων παίρνουν επιδόματα είναι λόγω πλήρους ανέχειας είναι γυναίκες. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Λάμπερτ από τους Πράσινους. Ο κύριος Μαραγκάλ, δεν είναι εδώ ο κύριος Λάμπερτ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ας μιλήσουμε για την Καταλωνία, δηλαδή για την Ευρώπη. Στην Καταλωνία αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξαιρετική διαδικασία αυτοδιάθεσης, ειρηνική και υψηλής δημοκρατικής ποιότητας. 2,3 εκατομμύρια ψήφοι το Νοέμβριο, 2 εκατομμύρια συμμετέχοντες το Σεπτέμβριο, 1,5 εκατομμύρια υπογραφές δήλωσης προς αυτή την κατεύθυνση. Ξανά και ξανά αρνείται ε, το Ισπανικό κράτος να ξεκινήσει διάλογο και να τον συνεχίσει και δεν τηρείται τους ίδιους, δεν τηρεί τους ίδιους κανόνες το rule of law, το κράτος δικαίου που ε, ζητούμε εμείς από οποιαδήποτε άλλη χώρα εάν πρόκειται να προσχωρήσει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον νόμο το καταλανικό για την εξωτερική δράση. Αναστάλθηκε η θέση ενός ε, δικαστή γιατί είχε ουσιαστικά πολιτικές θέσεις. Δηλαδή το καταργήθηκε από τη θέση του γιατί ε, δεν άρεσαν οι απόψεις τους. Επίσης καθαίρεσε το Ισπανικό κράτος τον Καταλανό διαμεσολαβητή. Ombudsman. Η Καταλωνία είναι μέρος της καλύτερης ευρωπαϊκής ελπίδας. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους ακραίους εθνικισμούς. Αντίθετα, ακραίο εθνικισμό επιδεικνύει το Ισπανικό κράτος. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αντιλαμβάνομαι ε, το θέμα με την Καταλωνία, αλλά ε, συγγνώμη σας διάκοψα, αλλά περάστε το χρονικό όριο. Ευχαριστώ πολύ, Ρόζα Νταμάτο. Ω μέλο τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη, θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για τα 300 προγραμμάτα στην Περιφερειακή Ανάπτυξη που χρειάζονται αναθεώρηση ώστε να μην χαθούν οι πόροι του 2014 Χρειάζεται λοιπόν αναθεώρηση του πολιετούς ε, πλαισίου που θα εξεταστεί σε αυτή την αίθουσα ε, στο εγγύς μέλλον για να αποφύγουμε παρόμοια προβλήματα στην επόμενη προγραμματική περίοδο επιθυμώ συνεργασία καλύτερη μεταξύ κρατών μελών Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και περιφερειακών και τοπικών αρχών η διαχείριση αυτή θα πρέπει να γίνεται από κοινού στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ωστόσο πρέπει να εκφράσω με επικρία ότι στη χώρα μου εδώ και δεκαετίες υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικότερα στις περιοχές του Νότου, οπότε ζητώ ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί ώστε να μην έχουν τα προβλήματα αυτά πάντα οι ίδιες περιοχές. Ευχαριστούμε. Φραντς Όμπρεμαγερ, ε, μην γεγραμμένος και ζητώ πάλι συγγνώμη για αυτό που συνέβη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της Αφρικής. Ξέρετε ότι υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη και οι οποίοι είναι μέλη Ισλαμιστικών κινημάτων. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί καθότι τα κύματα αυτά αυξάνονται και με τον ίδιο τρόπο βάζουμε και μια ορολογιακή βόμβα του Ισλαμισμού. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές στηρίζονται από θεσμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθότι πρόεδροι ιδρυμάτων και πολύ γνωστών φορέων καλούν και υποστηρίζουν πολλές φορές τέτοια κινήματα. Θα πρέπει να είμαστε ίσως πιο προσεκτικοί, να ασκήσουμε μια λίγο πιο αυστηρή κριτική σε αυτά τα ισλαμιστικά κινήματα, στον Ισλαμισμό, καθότι κινδυνεύουμε να μπουν από την πίσω πόρτα στην Ευρώπη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν δεν είμαστε προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Ε, ο Τομάς Tomasz Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή επικαλείται δικαιώματα κάθε είδους και πολλές φορές αγνοούμε το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Βλέπουμε ότι αυτό δεν το επικαλούνται πολλοί και πολλοί ξέρουμε παραδείγματα κατεστραμμένων οικογενειών, γυναικών παραδείγματος χάρη, οι οποίες δεν θέλουν σήμερα να αναφέρουν ποιος είναι ο πατέρας των παιδιών τους. Αρνούνται δηλαδή στους ε, ε, πατέρες το δικαίωμα να αναγνωρίσουν τα παιδιά τους και να ζήσουν και να παρακολουθήσουν την ε, ανατροφή τους. Πιστεύω ότι ένας άνδρας ο οποίος δεν μπορεί να αποδείξει την πατρότητά του είναι ένα δικαίωμα που του στερείται το οποίο επίσης θα πρέπει να επικαλεστούμε. Τα παιδιά, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρουν από πολιτικές σκοπιμότητες γι' αυτό οφείλουμε να τα ακούμε. σας μεταφέρω λοιπόν σύντομα μια επιστολή που μου έδωσαν τα παιδιά ενός δημοτικού σχολείου της Λευκοσία να σας μεταφέρω τις αγωνίες τους. είναι μόλις 8 χρονών. αναρωτιούνται γιατί να ζουν και να μεγαλώνουν σε μια μοιρασμένη πατρίδα όπου το 1 τρίτο να κατέχεται από ξένα τουρκικά στρατεύματα. αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν και αυτά τα παιδιά εντός της ευρώπης της ευρωπαϊκής ένωσης το δικαίωμα στην ελευθερία της πατρίδας τους αλλά και σε σχέση με την οικονομική κρίση αναρωτιούνται γιατί να μην έχουν φαγητό να φάνε και ρούχα να φορέσουν γιατί να υπάρχουν παιδιά δυστυχισμένα στην πατρίδα μας εντός της ευρωπαϊκής ένωσης. οι μονόπλευρες πολιτικές λιτότητας φταίνε. και τελειώνουν με μια φράση και μια υπόδειξη για όλους μας σεβαστείτε την κύπρο είναι και αυτή μια χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ, Τσεκοφσκή, από το ΕΣΥΑΡ. παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το 2008 έφταναν ε, ρωσικά αρμάτα ε, στη Γεωργία ε, και σήμερα λέμε ε, η Γεωργία και με ε, η Ουκρανία και μετά σύντομα θα είναι και η Πολωνία. Ξέρετε, η Ρωσία υπό τον Πούτιν ε, υλοποιεί αυτό το σενάριο. Το σενάριο σήμερα είναι η Ουκρανία. Και να δούμε τι έπεται. Ας ακούσουμε τον Ποροσέγκο που είπε ότι η πραγματική φιλοδοξία της Ρωσίας πηγαίνει πέραν της Ουκρανίας. Προσοχή, η ρωσική αυτοκρατορία που έχει χτίσει ο Πούτιν δεν τελειώνει στην Ουκρανία, ούτε καν στην Πολωνία. Μπορεί να φτάσει μέχρι το Βερολίνο. Θέλω λοιπόν να μας απασχολήσει, να απασχολήσει τους Γερμανούς πολιτικούς αυτός ο προβληματισμός. βάλει από το Uh, Ευχαριστώ. Τον Απρίλιο του 2016 η Ιρλανδία θα ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία τρεις νέες οδηγίες για τις κρατικές προμήθειες και τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι θετικό εργαλείο για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων, η αηφόρος ανάπτυξη και ε, να επιτευχθούν κοινωνικοί στόχοι όπως είναι ε, τα δημοσιονομικά. Ε, θέλουμε να έχουμε προβλέψεις για το περιβάλλον, για τις εργασιακές σχέσεις και όλα αυτά να αναφέρονται καθ' τη διάρκεια της ε, ε, διαδικασίας για τις κρατικές προμήθειες και συμβάσεις. Θα πρέπει πάντοτε να τηρούνται τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Η Ιρλανδία είναι η δεύτερη στον ΟΣΑ από πλευράς χαμηλών μισθών. Οι γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτες και αυτά πρέπει να τα γνωρίζουμε. Δεν θα πρέπει να συρρυκνώσουμε τις υπηρεσίες και θα πρέπει να παραμείνουν διάφορες υπηρεσίες σε κρατικό έλεγχο. Θα πρέπει να προστατευτούν και η τοπική αυτοδιοίκηση και δεν θα πρέπει να περάσουμε σε υπεργολαβίες και διαγωνισμούς ε, τέτοιου είδους για δημόσιες υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Η Τζούλια Μόη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, με εκπλήσει ότι εν ώψη της εκθέσης του Μιλάνου έγιναν εξαιρέσεις για εισαγωγές διατροφικών προϊόντων από τρίτες χώρες ενώ θα παραμείνουν κλειστές οι δυνατότητες μεταφοράς δικών μας προϊόντων. Έχουμε καταπληκτικά προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να ενδιαφέρουν όλους μας για αυτό το σημείο. Πολλές φορές έγινε η έκκληση προς την Κομισιόν για να μην γίνει αυτή η ντροπιαστική πράξη που πλήττει τους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς της Αρδενίας, Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους τοπικούς ε, πολιτικούς της Αρδενίας και τα κόμματα από το 1978 μέχρι σήμερα, δηλαδή σε μια περίοδο πάνω των 30 ετών, αντί να λύσουν το πρόβλημα, μόνο φωνάζουν και κάνουν το μόνο που γνωρίζουν να, αυξήνουν, να αυξάνουν τους δικούς τους παρασιτικούς μισθούς τους οποίους πληρώνουν οι ε, κάτοικοι της Αρδενίας. Να τους ευχαριστήσουμε σήμερα που πολλοί παραγωγικοί τομεί τη Ιταλία είχαν μια τεράστια ευκαιρία προώθηση τη εικόνα των προϊόντων μα. Η Expo 2015 είχε γεννηθεί ε, με κακούς ιονούς αλλά ελπίζω να μην καταλήξει να είναι ένα άντρο ε, ένας χώρος απάτης ευχαριστούμε ο κύριος ε, Λευτέρης Χριστοφόρου Κύριε Πρόεδρε είμαι υποχρεωμένο σήμερα να θέσω ενώπιον του Κοινοβουλίου του Ευρωκοινοβουλίου ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με την Κυπριακή ναυτιλία αλλά κατ' επέκταση με την Ευρωπαϊκή ναυτιλία εδώ και χρόνια η Τουρκία με πειρατικό παράνομο αυθαίρετο και κοινικό τρόπο επέβαλε ναυτικό εμπάρκο στα πλοία που φέρουν την κυπριακή σημαία και κατ' επέκταση επέβαλε εμπάρκο στα ευρωπαϊκά πλοία. είναι απαράδεκτο και αδιανόητο η τουρκία να παραμένει ανενόχλητη και ατιμόρυτη να παραβιάζει το πρωτόκολλο της άγκυρας που ήδη υπέγραψε και ουσιαστικά όφιλε μέχρι σήμερα να αναγνωρίσει την κυπριακή δημοκρατία και να ανοίξει τα λιμάνια και τους εθέρες και ουσιαστικά να προσβάλλει και να προκαλεί την ίδια την ευρωπαϊκή ένωση. εμείς ως κύπρος υφιστάμεθα τεράστιο ναυτιλιακό και οικονομικό κόστος. αυτό το κόστος το υφίσταται και η ίδια ευρωπαϊκή ένωση και η ίδια ευρωπαϊκή ένωση την ίδια τη στιγμή που υφίσταται κόστο από χώρα υποένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση που είναι η τουρκία ουσιαστικά ανέχεται και παρέχει και προενταξιακή βοήθεια στην τουρκία. φανταστήκατε κύριε πρόεδρε τελειώνοντας σε αυτό το ευρωκοινοβούλιο τι θα γινόταν ή στην ευρωπαϊκή επιτροπή εάν η τουρκία απαγόρευε σε πλοία με βρετανική γαλλική ή ιταλική σημαία να μπαίνουν στα λιμάνια της. Ευχαριστώ. Πάνι Μάρια Ευχαριστώ κυρία Γραπίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Φεβρουάριο φέτος της 23 η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων ανέφερε τη συμπερίληψη της Ρουμανίας ε, στη διαδικασία μακροοικονομικών ισορροπιών ε, ήταν ασαφής η λογική, η εφαρμογή αυτής της παρακολούθησης απαιτεί σύμφωνα με την νομοθεσία την υπέρβαση ορισμένων κατοφλίων όσον αφορά του ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών ε, της συναλλαγματικών ισοτιμιών του ενωπημένου χρέους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κανένας από αυτούς τους δείκτες δεν έχει φτάσει στα κρίσιμα κατόφλια στη χώρα μου ώστε να συμπεριληφθεί στη διαδικασία παρακολούθησης. Η Ρουμανία περνάει το τέταρτο έτος οικονομικής ανάπτυξης, έχει σταθερό η συναλλαγματική ισοτιμία, αύξηση των εξαγωγών, καμία πτώχευση στον τραπεζικό τομέα και οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις βρισκόνται καθοδόν. Μπορούμε να εξαγούμε το συμπέρασμα λοιπόν ότι η απόφαση της Ρουμανίας να μην επεκτείνει τη συμφωνία της με το δουνό του συμπεριλαμβάνεται. Ε, θεωρώ ότι είναι λανθασμένη η κίνηση αυτή και θεωρώ ότι η Κομισιόν έχει την υποχρέωση να παράσχει συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Για ποιο λόγο συμπεριέλαβε τη Ρουμανία σε αυτή τη λίστα, ε, πράγμα που επηρεάζει την αξιοπιστία τη Ρουμανία προ του επενδυτέ τη. Ε, ευχαριστώ, ο κύριο Φιλιππλόσο. Παρακαλώ. Με εγγεγραμμένο. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται ότι και άλλες χώρες θα μπορέσουν να υποφεληθούν από την οικονομική αυτή ενώ άλλες χώρες πλήττονται και υποφέρουν. Βλέπουμε ότι για τα 11 δισεκατομμύρια προϋπολογισμό για την διεύρυνση και χώρες ταυτόχρονα που προετοιμάζουν την προσχώρησή τους. Βλέπουμε ότι σήμερα πάνω από 5 δισεκατομμύρια έχουν διατεθεί προς αυτό το σκοπό. Σήμερα όμως εγώ πήρα το λόγο για να μιλήσω για έναν τομέα που χρηματοδοτείται και στηρίζει αυτό το εργαλείο. Ο εξυγχρονισμός της γεωργίας αυτών των χωρών που πρόκειται να προσχωρήσουν και που την ίδια ώρα τα προϊόντα τους ε, ανταγωνίζονται με ακόμα έναν τρόπο τα δικά μας προϊόντα και εδώ αναφέρομαι στην χώρα μου, στη Γαλλία, όπου πάρα πολλοί αγρότες σήμερα υποφέρουν. Ευχαριστώ. Κάρλος Τρουγέης, από το ΕΛΚ. Την περασμένη εβδομάδα πέρασαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ορισμένοι συγγενείς των εγκληματιών της ΕΤΑ, της τρομοκρατικής οργάνωσης και είδαμε ότι χρησιμοποιούνται οι συγγενείς αυτοί για να νοποιημοποιήσουν την τρομοκρατική οργάνωση. Οι συγγενείς αυτοί δεν θέλουν να ζητήσουν συγγνώμη για τις δολοφονίες που έχουν διαπράξει τα μέλη της οικογένειά τους που είναι, βρίσκονται στην φυλακή. Και ξέρετε, η Ετσεράτη είναι επίσης ε, ε, τρομοκρατική οργάνωση και είναι παρακλάδι της ΕΤΑ. Ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί προσπάθησε να κοροϊδέψει κάποιους τελικά και να τους οδηγήσει σε λάθος ε, μονοπάτια. Θέλουν να φαίνονται θύματα αλλά είναι ιδίμιοι. και μάλιστα η διαφορά είναι πια μεταξύ των οπαδών και φίλων της ΕΤΑ μπορεί κανείς να επισκεφθεί ε, τους δολοφόνους. Οι συγγενείς και φίλοι των ε, τρομοκρατών μπορούν να τους επισκεφθούν. Οι συγγενείς των θυμάτων όμως μόνο τους τάφους μπορούν να επισκεφθούν. Και αυτή είναι η πραγματική αλήθεια σε αυτή τη ιστορία. Και μόνο αυτό γίνεται με την Ετσεράτ, με αυτή την οργάνωση τρομοκρατική που είναι παρακλάδη της ΕΤΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Σενάλαβα παρακαλώ από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κόστος των τροφίμων ε, είναι το 40% του οικογενειακού προϋπολογισμού. Από 20% έως 40% κυμαίνεται. Έχει αντίκτυπο σε κάθε καταναλωτή, αλλά έχει και τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομία. Ξέρετε πολλοί αγρότες, παραγωγή τροφίμων εν γέννη, θεωρούν ότι τα περιθώρια κέρδους του λιανεμπορίου είναι τεράστια. Έχουν διπλασιαστεί από το 2009 μέχρι σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είχε εξετάσει αυτό το θέμα πριν από πολλά χρόνια, όμως συνεχίζουμε να μην γνωρίζουμε ε, ποια είναι τα περιθώρια κέρδους ε, του λιανεπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν ε, και διαμορφώνουν τη τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Αυτό θα ωφελήσει όλους και την τροφική αλυσίδα και τους καταναλωτές. Ο κύριος Κέλλη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω συμμετάσχει σε μια εκστρατεία και συμμετέχω σε μια εκστρατεία προώθησης της μητρικής γλώσσας είναι η Ιρλανδική Εβδομάδα ε, Ιρλανδικής Γλώσσας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα εδώ, διότι υπάρχει υπηρεσία δερμηνίας ε, και οι δερμηνείς μεταφράζουν τα λεγόμενά μου. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα δημιουργηθεί ε, και, απασχόληση. Θα υπάρξουν θέσεις απασχόλησης για μεταφραστές, για διερμηνείς, για τη μετάφραση των ευρωπαϊκών εγγράφων. Την επομένη εβδομάδα, ξέρετε, είναι η μέρα του Αργίου Πατρικίου, που είναι εθνική μας εορτή και θα οργανώσουμε ε, μία σχετική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα λοιπόν, αντί να πω στη γυναικιά μας, αντί ε, στην υγειά σας ή η καλή σας όρεξη, θα ήθελα να πω σλάνισε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και σλάνισε στα Ιρλανδικά. Thank you very much It was really nice. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ευχαριστώ. Κύριε Ραλέγγ από τους σοσιαλιστές, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το Μπιμίος είναι από, από τα μεγαλύτερα μουσεία, ανοιχτά μουσεία με πολλές χιλιάδες ε, επισκέπτες το χρόνο. Είναι σημαντικός εργοδότης ε, στη βορειοανατολική Αγγλία από που προέρχομαι. Η βιομηχανία του, ο τομέας του πολιτισμού αφορά χιλιάδες θέσεις εργασίας ε, ε, και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και πολλές ε, μπενεκτούς ομάδες και αποτελεί στοιχείο κλειδί της οικονομίας μας η βορειοανατολική συνεργασία στον τομέα του πολιτισμού ε, χρησιμοποιεί κονδύλια από την Ευρώπη τα οποία όμως έχει μπλοκάρει η Βρετανική κυβέρνηση για τον τομέα του πολιτισμού αγνοώντας τα κοινωνικονομικά ωφέλη που προσφέρει η Ευρώπη για τον τομέα του πολιτισμού σε εποχές όπου οι περιοχές μας δεν έχουν περιθώριο να απορρίψουν δυνατότητες δημιουργίας, ε, ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βίνκλερ. Eh, eh, Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και τρεις εβδομάδες μάλλον πριν από τρεις εβδομάδες κάποιοι άγνωστοι κατέστρεψαν τα μνήματα 13 ηρώων της Ουγγαρίας, της χώρας μου. Πρόκειται για μνημεία από την Ουγγαρία και την Ρουμανία. Η γαλλογερμανική φιλία είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει σήμερα να μεταβληθεί σε σύγκρουση και σε διαμάχη και το ίδιο πρέπει να γίνει και στη δική μας περιοχή. Πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτά τα ακραία κινήματα και το φανατισμό. Πρόεδρος. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, από τους Σοσιαλιστές, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπήρξαν πολλές πλημμύρες στο κέντρο της Ευρώπης πριν από χρόνια και η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη είναι αυτή που δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και Προστασίας έναντι των φυσικών καταστροφών ε, και έχει πρικοδοτηθεί με 500 εκατομμύρια ευρώ. Και εμείς ζηλέψαμε πάρα πολύ γιατί στην Αραγωνία υπάρχει ο ποταμός Εύρος. Είναι ένας πολύ πλούσιος ποταμός που έχει πολύ έφορα εδάφη γύρω του πλημμύρισε και καταστράφηκαν πάρα πολλές καλλιέργειες. Βρήκαν το θάνατο 10.000 ζώα, 28.000 εκτάρια επλήγησαν. Είχαμε τεράστιες πλημμύρες, ε, καταστροφή θερμοκηπίων. Ήταν μια πολύ άσχημη κατάσταση σε γενικές γραμμές. Η περιφερειακή κυβέρνηση και η εθνική κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος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 να βρίσκεται στο επίκεντρο ε, των όλων των πολιτικών μας. Είναι μια ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα. Είναι μια ευκαιρία για την έρευνα, για την, ε, ε, ε τους επαγγελματίες φροντίδας και υγείας. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ενθαρρύνουν την οικονομία μας. Είναι κίνητρο για να αναθεωρήσουμε το, το, τα εθνικά συστήματα υγείας στις χώρες μέλη η τρίτη ηλικία στην Ευρώπη θα πρέπει να έχει αυτονομία, αυτάρκεια και να μπορεί να ζει ε, με υψηλή ποιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δράκης, παρακαλώ. Στις 3 Μαρτίου στην Ιταλική τηλεόραση η κυρία Διανά Παύλοβιτς, η στη ρατσιστική επίθεση από τον Τζαλούκα Μπονάνο Ιταλό βουλευτή εγώ ως, Ρωμαίος βουλευτή, ως Ρουμάνος βουλευτής ως πολίτης Ρουμανίας και πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορώ να δεχθώ τέτοια δημόσια συμπεριφορά διότι η πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκω οι σοσιαλιστές σε 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να με υποστηρίξει για να γίνω μέλος αυτού εδώ του θεσμού αλλά δεν υποστηρίζει την καταγγελία αυτής της συμπεριφοράς αν έχετε αμφιβολίες για το ποιοι είναι και για το, ε, ε, σε ποιους αναφέρομαι να σας υπενθυμίσω όποιος έχει ρατσιστική στάση να θυμάται τον Τζάλο Καμπονάνο ως ε, μέλος του Κοινοβουλίου ότι αυτό θεσμικό χρόνο δεν επιτρέπει τέτοια δημόσια συμπεριφορά η κατάσταση ε, είναι τέτοια πρέπει να επιβάλλεται κυρώσει κατά τέτοιων συμπεριφορών. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, κάνω έκκληση προς το Κοινοβούλιο να λάβει δημοσίως στάση ε, και να κατηγορεί τέτοιες συμπεριφορές όπου εμφανίζονται. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιβάνα Μαλέτητσα από το ΕΛΚΑ Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρη δράση γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές οι πολίτες της Ευρώπης είναι θύματα. Το 2014 βλέπαμε ανθρώπους να ζουν σε κοντέινερ, σε άθλιες συνθήκες και θα πρέπει σαφώς να υποστηρίξουμε τις ε, οργανώσεις αυτές που τους στηρίζουν. Βλέπουμε επίσης ότι οι εργοδότες έχουν μια πάρα πολύ απαράδεκτη συμπεριφορά προς αυτούς τους, τις ευάλωτες κατηγορίες που πολλές φορές είναι και πολλοί νέοι άνθρωποι. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτούς τους πολίτες, να τους εγγυηθούμε ασφάλεια, αλληλεγγύη και οι κανόνες καλής οικονομικής διακυβέρνησης να ισχύσουν και για αυτούς. Ο τελευταίος ομιλητής είναι η Έστερ Καρσιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Ισπανικής Αντιπροσωπείας του Λαϊκού Κόμματος των κυρίων Ντεναβάρα και Λόπεθ Φοντανιέρ που δεν μπόρεσαν να μιλήσουν και εμείς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας ε, για, προς τους πολίτες της Αραγωνίας που διαβιούν κοντά στον ποταμό Εύρο ο οποίος πλημμύρισε τέσσερις φορές αυτή την εβδομάδα ήταν τεράστια φυσική καταστροφή ε, μεγάλο πλήγμα για χιλιάδες οικογένειες που ζουν από την κτηνοτροφία και τη γεωργία. Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε τις αυτόνομες κοινότητες της Λαριόχα και της Αραγωνίας για τη βοήθεια που προσφέρουν και περιμένουμε να υπάρξει βασιλικό ε, διάταγμα ε, της Ισπανίας για να υπάρξει αποζημίωση των πληγέντων και αν δεν είχαμε 7 χρόνια σοσιαλιστική κυβέρνηση θα είχαμε προλάβει και θα είχαμε μπορέσει να κάνουμε τα έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για να προλαμβάνονται τέτοιου είδους πλημμύρες. Ε, σε κάθε περίπτωση εμείς θα το πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή στη συζήτηση. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για την παρουσία της εδώ. Κυρίες και κύριοι, κυρίσω το πέρασε τη συνεδρίασής μας. Συνεχίζεται η Ολομέλεια αύριο το πρωί στις 8.30 μέχρι τις 2 και μετά από τις 3 μέχρι τις 11. Την ημερήσια διάταξη θα τη βρείτε στη διαδικτυακή.